εξ ονόματος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ευρωπαίων Δημοκρατών δίνω το λόγο στον κύριο Ζωζεφ Ντόλ παρακαλώ. Πρόεδρε. Κύριοι Πρόεδροι του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε γιατί θεωρούμε εκ μέρους της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ότι ο κύριος Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόσο και τα μέλη της Επιτροπής μαζί με το ε, της Επιτροπής Συλλογικό Όργανο θα είναι κατάλληλοι για να επιτελέσουν το έργο για το οποίο έχει προβλεφθεί ο διορισμός τους. Γιατί έχουμε να κάνουμε, ύστερα από τόσα δεκαετίες ευρωπαϊκού ολοκληρώματος, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ε, με ένα πολύ μεγάλο αγώνα, με μια μεγάλη προσπάθεια γιατί πρέπει να διασώσουμε το ευρώ, το ευρώ το οποίο έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σταματήσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ... Έχετε το χρόνο, έχετε ε, εκμεταλλευτεί και εσείς τις ευκαιρίες που σας έδωσε το ευρώ, κυρίες και κύριοι φίλοι. Σε ποια κατάσταση ήταν, δεν υπήρχαν οι σταθεροποιητές της ε, αλληλεγγύης που πολλές φορές θεωρήθηκαν βαρύδι στις οικονομίες μας που όμως συνέβαλαν τόσο πολύ στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού μοντέλου, ενός μοντέλου το οποίο είναι ελκυστικό, το οποίο μιμούνται και άλλοι και το οποίο όλοι, στο οποίο είμαστε όλοι προεδεμένοι με, με αφοσίωση, που όμως πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, γιατί ο κόσμος πλέον είναι πολυπολικός, όχι όπως το φανταζόμασταν όμως πολυπολικό, δηλαδή ειρηνικό και πολυπλευρό, αλλά πολυπολικός μέσα από τον ανταγωνισμό, μέσα από έναν αγώνα έστω ειρηνικό, αλλά σκληρό, σκληρότατο για την επιβολή του μοντέλου του ενός πάνω στους άλλους. Έτσι λοιπόν αυτός ο κόσμος, το ευρώ το δικό μας, το οποίο έχει τόσα ε, πλέον εκτήματα, η Ευρώπη αυτή η οποία είναι υπόδειγμα ε, για την ε, προαγωγή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για όλα αυτά τα θετικά πράγματα πρέπει να παραμείνει ελκυστική και ταυτόχρονα σε θέση ανταγωνιστική. Και σε αυτό πιστεύω ότι θα αγωνιστεί η νέα Επιτροπή. Όλοι βεβαίως γνωρίζουμε ποιες είναι οι μεγάλες ε, δυσκολίες, η δημογραφία χαμηλή, ο προϋπολογισμός, ο πληθωρισμός το εξωτερικά χρέη, το ευρωπαϊκό νόμισμα όμως μπορεί να αποτελέσει ε, εχέγγυο και για την επιστηστική βοήθεια, για τη γεωργία δηλαδή και για την, ε, και διατράνωση της βιομηχανίας μας και για την παρουσία της Ευρώπης στις διεθνείς αγορές και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτελέσει αυτό το έργο και περιμένω ότι η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, προαγάγει τα συμφέροντα της Ευρώπης, ότι θα διατρανώσει τις θέσεις μας ε, και την παρουσία μας στη συνεργασία με τους εταίρους μας και ότι θα είναι πάντα παρούσα στους μεγάλους αγώνες. Κυρίες και κύριοι Επίτροπε, εσείς μαζί με εμά, ε, μαζί με το Συμβούλιο, καλούμεθα όλοι μαζί να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά και γι' αυτό θα πρέπει να διαρρήξουμε τα ταμπού της φορολογίας και των κοινωνικών. Δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να ε, ισχυρίζονται πλέον ότι βρίσκονται στο απειρόβλητο αυτές οι αρμοδιότητες και έξω από την κοινή κοινοτική δράση. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να, να διπλασιάσουμε, να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας τι εξωτερικές προκλήσεις και για την ασφάλεια και για τις κοινωνικές ε, προδιαγραφές και για τις βιομηχανικές προδιαγραφές και για τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Η Ευρώπη θα πρέπει να προασπιστεί των αξιών, τη ειρήνης, τη ευημερία των πολιτών τη. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ένα παράγοντα παγκόσμιο και όχι μόνο ένας χώρος ευημερία και δικαιωμάτων. Δεν μπορεί η Ευρώπη να απεμπολίσει τα μέσα ε, που της επιτρέπουν να εξασφαλίσει περισσότερη ισχύ και πιστεύει η ομάδα μας ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το πεδίο να αγωνιστεί ιδιαίτερως. Αν το κάνει αυτό και είμαι βέβαιο ότι θα το πράξει, το ΕΛΚ θα είναι πάντοτε στο πλευρό της. Πρόεδρε Ζωζέ Μπαρόσο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σας εκφράζει την εμπιστοσύνη του και σας καλεί να αναλάβετε τι μεταρρυθμίσει με παρησία, με θάρρο, με όραμα για την ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή της ε, ε, πολιτικής Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντόρ. για την προοδευτική σοσιαλιστική ομάδα, ο Μάρτιν Σούλτ, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες την απόφαση αυτή δεν την έλαβαν ελαφρά την καρδία. Εδώ ψηφίσαμε πριν από πέντε μήνες για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τότε δεν δώσαμε την εμπιστοσύνη μας, αλλά πήρε πλειοψηφία και με βάση αυτή την πλειοψηφία που δυστυχώ εξαρτάται από άτομα που δεν ήταν υπέρ τη συνθήκη Λισαβόνα, με βάση αυτή την πλειοψηφία μα παρουσίασε ένα σώμα επιτρόπων. Σήμερα πρόκειται αυτό το σώμα των επιτρόπων να αξιολογηθεί από εμά, να αποτιμηθεί. Πρέπει να το αποτιμήσουμε και να το αξιολογήσουμε. Δύο δυνατότητε έχουμε. Μπορούμε να διχαστούμε στου αριστερού και στου δεξιού και να πούμε βρισκόμαστε σε μια ιδεολογική αντιπαράθεση δεξί και αριστερή, και έτσι θα ψηφίσουμε. Αυτό είναι η μία δυνατότητα. Αλλά έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρώπη. Εμείς σε αυτή την Ευρωβουλή δεν έχουμε πλειοψηφία. Το ΕΛΚ σε αυτή την Ευρωβουλή δεν έχει πλειοψηφία. Οι Άλντε δεν έχουν πλειοψηφία. Η Ευρώπη δεν είναι μόρφωμα όπου κάποια πολιτική δύναμη αυτή μόνη τη μπορεί να δημιουργήσει τα πράγματα και να πει έτσι ακριβώ κομμένο και ραμμένο θα είναι το κοστούμι τη Ευρώπη εφ' εξής. Η Ευρώπη είναι διαρκή συμβιβασμό. Αυτό κάνει καμιά φορά τόσο δυσλειτουργική, τόσο δυσνόητη την Ευρώπη. Αλλά καλύτερο είναι ο συμβιβασμό που οδηγεί σε επιτυχίε και μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη από την ιδεολογική αντιπαράθεση που στο τέλο χωρί κανένα πρακτικό αποτέλεσμα οδηγεί οδηγεί σε εξάντληση. Και γι' αυτό για μας είναι δύσκολο να αποτιμήσουμε απόλυτα σωστά. Φυσικά έχουν ολοκληρωθεί τα πράγματα και θα έκαναν μεγαλύτερη ευχαρίστηση με τους συναδέφους άλλων τερίγων να μπορούμε επί των θεμάτων αρχίσει να αντιτιθέμεθα. Όμως χρειάζεται χειροπιαστά αποτελέσματα η Ευρώπη. Γι' αυτό θέσαμε το ερώτημα τι μπορούμε εμείς ως σοσιαλδημοκράτες, ως σοσιαλιστές και δημοκράτες να απαιτήσουμε και τι μπορούμε να πετύχουμε και να περάσουμε. Και καθορίσαμε κάποια κριτήρια. Ένα κριτήριο ήταν ότι θέλαμε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανώτατο επίπεδο την πολιτική δύναμη που είναι η δεύτερη δύναμη στην Ευρώπη να την εκπροσωπούμε. Και γι' αυτό την είπα το εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, καταφέραμε να πετύχουμε αυτό το αξίωμα. Και θέλω να πω για την κάθε Άστον που έχει αυτό το αξίωμα. Η κάθε Άστον πρέπει σε αυτή την Ευρωβουλή, κυρίες και κύριοι, όχι να ακούει ότι είναι λέει κομμουνίστρια από κάποιον που στη Γαλλία έχει καταδικαστεί από δικαστήρια ως αρνητής του ολοκαυτώματος. Η κάθε άστον έχει την πλήρη εμπιστοσύνη μας, Είναι εμπιστοσύνη όλων μας. Εμείς θέσαμε το ερώτημα και είπαμε μπορούμε να αποτιμήσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις σαν ένα ρυθμιστικό μηχανισμό στον, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να θεσπίσουμε αυτή την λειτουργία. Για μας το ερώτημα ήταν μέτρα, π.χ. όπως η Οδηγία Περιπαροχής Υπηρεσιών στο παρελθόν, αν μπορούν να δρομολογηθούν και να προχωρήσουν. Θέλαμε ένα μηχανισμό που θα εξετάζει και θα αποτιμά ότι κάθε μέτρο που θα υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγχεται προτού ληφθεί για τις επιπτώσεις της, για τα συστήματα των κοινωνικών ασφαλίσεων στα κράτη-μέλη. Αυτό κατοχυρώθηκε τώρα πλέον. Θέλαμε και για μας αυτό είναι ποιοτικό άλμα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Τα νομοθετικά ψηφίσματα αυτής της Ευρωβουλής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνονται και να υιοθετούνται και να αναλαμβάνει η νομοθετική πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω αυτών. Αυτό είναι τεράστια πρόοδο. Διότι το δυστυχώ μη υπάρχον, μη υφιστάμενο δίκαιο πρωτοβουλία, δικαίωμα πρωτοβουλία του Ευρωκοινοβουλίου με αυτόν τον τρόπο μεταφράζεται χειροπιαστά. Αυτό είναι πρόοδο για μα, μεγάλη πρόοδο. Και τέλο θέλαμε να πετύχουμε ότι η δύναμη που έχουμε σε αυτό το κοινοβούλιο σαν δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη που δεν καταφέρνει να πετύχει μια ε, ειδική πλειοψηφία να μπορεί αυτή η δύναμη να μεταφράζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρει από του επτά αντιπροέδρου είναι σοσιαλδημοκράτε. Εκεί υπήρξε ανταπόκριση λοιπόν. Και πολλά πολλές επιφυλάξεις διατυπώσαμε τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες και σήμερα το πρωί πάλι στις συζητήσεις μας. Αφήσαμε να εννοηθούν να ακουστούν οι επιφυλάξεις που έχουμε ακόμα στην ε, αποτίμηση αυτών των επιφυλάξεων και στις προόδους που επιτύχαμε αποφασίσαμε να εκφράσουμε σε εσά την εμπιστοσύνη μας για τα επόμενα αυτά πέντε χρόνια της θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν λέω σε εσά, αυτό ισχύει για το σώμα των επιτρόπων συλλογικά γυναικών και ανδρών μπορείτε να βασίζεστε στην υποστήριξή μας. Αν πάρετε στα σοβαρά αυτές τις συστάσεις που σας διατύπωσα, είτε θα είναι κοινωνική αυτή η Ευρώπη ή θα αποτύχει. Αυτό είναι κοινή ευθύνη όλων μας. Να μεριμνήσουμε ότι θα είναι κοινωνική αυτή η Ευρώπη. Η σοσιαλδημοκρατική ομάδα θα εκφράσει την εμπιστοσύνη της σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκίφερ Χοφστάτ τώρα. Ε, εκπρόσωπος, ε, εκπρόσωπος των Φιλελευθέρων. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα μου θα υποστηρίξει την ε, νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Συμμαχία των Φιλελευθέρων και των Δημοκρατών είναι μια υπεύθυνη ομάδα. Είναι μια υπεύθυνη ομάδα και πιστεύουμε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι τόσο κρίσιμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαίους πολίτες που χρειάζεται μια επιτροπή που να είναι σε θέση να ε, χέρι μιας ευρείας ε, υπερευρωπαϊκής υποστήριξης από πλευράς του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά θα είμαι και σαφής, Πρόεδρε. Η υποστήριξή μας είναι υπό όρους, πολύ περισσότερο από τα περασμένα πέντε χρόνια. Εμείς αναμένουμε η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποτελέσει την ατομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο θαραλέα, πιο φιλόδοξη και μια πιο ολοκληρωμένη οικονομική και κοινωνική προσέγγιση. Μια επιτροπή που θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι στην πρωτοπορία μια τέτοια στρατηγική που θα επιβάλλει στα κράτη-μέλη, θα τα αναγκάσει να κάνουν αυτό που οφείλουν να κάνουν. Και σίγουρα στην Ευρωζώνη θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πω υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μια πραγματική οικονομική, και μάλλον έναν πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό πυλώνα δίπλα στον νομισματικό. Τα, προβλήματα τη Ευρωζώνη σήμερα από αποτελούν την απόδειξη της αποτυχίας της αδύναμης προσέγγισης που ακολουθήσαμε στο παρελθόν τα τελευταία δέκα χρόνια με την υποτιθέμενο η μέθοδο ε, του ανοιχτού συντονισμού. Το ίδιο ισχύει και για άλλου τομεί. Στι κλιματικέ αλλαγέ, στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική πολιτική. Και η βασική υπόθεση πίσω από αυτήν την πιο τολμηρή προσέγγιση είναι ε, ότι στον πολυπολικό αυρενό κόσμο η Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο χωρίς να είναι πιο αποτελεσματική και χωρίς ε, περαιτέρω εμβάθυνση τη ολοκλήρωση της και μάλιστα στο εγγύ μέλλον. Αναμένουμε από εσά να αγκαλιάσετε αυτή την ε, προϋπόθεση, να μας προτείνετε σαφείς, σταθερές, φιλόδοξες προτάσεις σε όλους αυτούς τους ε, τομείς, καθώς και μεταρρυθμίσεις και ελπίζουμε ότι για να τα πετύχετε όλα αυτά θα χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα πρωτοβουλία σας στο πλήρες του δυναμικό. Σαφώς και μιλώ για ολόκληρη την Επιτροπή, για το σύνολο της Επιτροπής κύριε Πρόεδρε. Συνεργασία ως ένα σύνολο επιτρόπων, ως ένα ε, ε πολιτικό σώμα το οποίο θα προωθεί τις πολιτικές του. Μια ισχυρή κομισιόν είναι απαραίτητη. Η συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει νέα εργαλεία και έχει ενδυναμώσει και αυξήσει τις δυνατότητες δράσης μας. Και προς την κυρία Άστον να πω, σας ζητούμε, χρησιμοποιήστε τα αυτά τα εργαλεία. Χρησιμοποιούμε, θέλουμε περισσότερα από τον ε, είπα το εκπρόσωπό μας από ό,τι μέχρι τώρα. Ο ρόλος σας το απαιτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρειάζεται και το ζητά. Ε, εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες. Το δίδαγμα από την ΑΕΤ είναι ένα παράδειγμα. Ε, για να τοποθετήσετε γρήγορα την έκθεση για την ε, πολιτική προστασία ε, στο τραπέζι του Συμβουλίου για συζήτηση άμεσα για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς μας στόχους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Και τώρα, εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων, Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία, το λόγο έχει ο κύριος Δανιέλ Κονπεντίτ, πρόεδρος της ομάδας. Γιατί είστε τόσο εκνευρισμένοι, Σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν γίνεται συζήτηση εδώ. Έχουμε να κάνουμε μόνο με δηλώσει των αρχηγών των πολιτικών ομάδων. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων δεν ισχύει η διαδικασία της, του μπλε δελτίου. Δεν εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία. Δεν μπορείτε να αντιδράτε. Πρόκειται μόνο για δηλώσει των αρχηγών των πολιτικών ομάδων και γι' αυτό λόγο δεν λαμβάνω υπόψη τι αντιδράσει σα. Κύριε Κονβεντήτ. Κύριος Κολπεντίτ, μπορείς σε παρακαλώ να κλείσει το στόμα σου. Κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ομάδα των Πρασίνων δεν θα υπερψηφίσει την Επιτροπή. Και ταυτόχρονα υποβάλλουμε τις ιδέες μας, την ε, ε, τα οράματά μας για την Ευρώπη και την αποφασιστικότητά μας για αυτήν. Μην ισχυριστείτε κύριε Μπαρόσο ότι όποιος δεν ψηφίσει την Επιτροπή σας είναι κατά της Ευρώπης. Τέτοια παιχνίδια με εμά, του πράσινου Ευρώπης, δεν μπορείτε να τα παίξετε. Με τους άλλους ίσως. Εμεί σα προτείνουμε συνεργασία χωρί αντιρρήσει, χωρί χωρίς αντιρρήσει. Εάν θέλετε να προχωρήσετε σε μια ευρωπαϊκή φορολογία, εάν θέλετε ιδίου σπόρους Ευρωπαϊκού, ναι, θα σταθούμε δίπλα σα κατά τη οικονομική επικυριαρχίας των κρατών και τα ε, κατανομάζω είτε είναι η Γερμανία είτε είναι η Γαλλία, αυτά εμεί θα σταθούμε στο πλευρό σα. Και αν θέλετε να είστε εσεί οι εγγυητέ, ο εγγυητή των συνθήκων, σήμερα παραδείγματι, διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο για την... Ε, επιστροφή ε, των προσφύγων στη Λιβύη γίνεται αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η νομική βάση μας λέει η Επιτροπή με ποια νομική βάση θα, γίνει αυτή, θα ληφθεί αυτή η απόφαση. Εσείς δεν λέτε τίποτα, εμείς λέμε ότι χρειάζεται συναπόφαση. Το Συμβούλιο μας λέει στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα ληφθεί η απόφαση για την, για την νομική βάση. Όχι λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση εγκαίρως για την νομική βάση αυτών των διαπραγματεύσεων. Και υπάρχουν μια σειρά παραδειγμάτων. Εάν θέλετε να προχωρήσετε, εάν θέλετε να επιδεινώσετε ακόμη περισσότερο το περιβάλλον, εάν θέλετε η Ευρώπη να περάσει περισσότερο αν θέλετε να αντιμετωπίσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ, αν θέλετε η Ευρώπη να πάει πιο μπροστά στα, στα τριπλ, στο τριπλό εικοσάρι, ε, αν θέλετε να πάμε πιο μπροστά ακόμη στη ρύθμιση των δημοσιονομικών μετά τη, και των χρηματοπιστωτικών συστημάτων μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, στο πλευρό σα θα είμαστε. Με πλήρη συνεργασία θα σταθούμε δίπλα σα. Εάν θέλετε μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προχωρήσετε περισσότερο για την προστασία τη Ευρώπη, ναι θα είμαστε στο πλευρό σα. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το κυπριακό πρόβλημα, ναι θα είμαστε στο πλευρό σα. Εάν θέλετε να σταματήσουμε επιπλέον επιτέλους ανοησίες όπως παλαβομάρες όπως ε, ε, το γεγονός ότι οι χώρες όπως η Ελλάδα δαπανούν 4,5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, για τέτοιους στόχους, ναι, θα είμαστε δίπλα σας ανεφόρον, θα σας, θα σας στηρίξουμε. Το είπα πολλές φορές και κύριε Μπαρόσο, μπορεί να σφάλουμε που σας ε, καταψηφίζουμε τώρα, την προηγούμενη φορά σφάλαμε ως προς την ψηφοφορία για τον κύριο Δήμα. Το ομολογούμε. Εάν λοιπόν εσείς ε, ε, αποδειχθείτε στο ύψος των περιστάσεων και όχι στο ύψος των όσων μας δηλώσατε σήμερα, θα είμαστε έτοιμοι να ομολογήσουμε ότι απατηθήκαμε, ότι σφάλαμε και θα είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε μια άλλη φορά. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο για ο κύριο Κίρκοπ εξ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών τη Ευρώπη. Ορισμένα κρατημέλη πιστεύουν ότι ο ορισμό ενό επιτρόπου είναι μια χρήσιμη ευκαιρία για την επίλυση κάποιου εσωτερικού προβλήματο ή για τη ρύθμιση ενό πολιτικού χρέου. Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν θα πρέπει να συγκεντρώνει του πιο ταλαντούχου ε, πολιτικού ηγέτε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανθρώπου με εμπειρία και ικανότητα για να αντιμετωπίσουν τι τεράστιε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Και μετά από ε, χρόνια θεσμική. Ε, ε, προχειρότητες ε, περιμένουμε αυτή τη στιγμή να υπάρξει μεγάλη συνεργασία. Θα πρέπει να μπορέσουμε να προωθήσουμε την έφραυτη οικονομική ανάκαμψη και να παίξει και ηγετικό ρόλο στην ενέργεια, στην ασφάλεια και στις κλιματικές αλλαγές και να προτείνει επίσης κεντρικές μεταρρυθμίσεις για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό καθώς και για πολλά από τα προγράμματα κλειδιά για τις δαπάνες. Και έχουμε βέβαια το σωστόν ηγέτη, κύριε Μπαρόζο, για να, προ, για να παροτρύνει ολόκληρη την Επιτροπή. Μια ατζέντα που εν γέννη υποστηρίζουμε. Κάθε μεμονωμένο κράτος θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειές του και να στείλει έναν ισχυρό υποψήφιο. Φυσικά και πρέπει να υποστηρίξει κάθε μέλος της ομάδας του. Αυτό και μόνο θα περιμέναμε από έναν ηγέτη στη θέση του και στην διοργάνωση αυτής της ομάδας, ε, αν και αμφισβητήσαμε κάποια χαρτοφυλάκια, προφανώς έκανε ό,τι μπορούσε με τα δεδομένα που είχε. Ορισμένοι υποψήφοι είναι πολύ καλοί και απέδωσαν πολύ καλά στις ακροάσεις. Ορισμένοι άλλοι είναι ε, μέτροι και δυσκολεύτηκαν. Εμείς βεβαίως ε, αν ε, εγκριθείτε θα, είμαστε, θα συνεργαστούμε στενά με όλους τους επιτρόπους και ελπίζουμε ότι θα εκπλαγούμε ευχάριστα. Αλλά ε, ετησίως θα σας ελέγχουμε. Πρόεδρε, πρόκειται για μια διαδικασία, μια διαδικασία που δεν μπορούμε να τη ολοκληρωτικά και γι' αυτούς τους λόγους οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές σήμερα θα πέσχουν από τις ψήφου. Ορισμένε ομάδε, κύριε Πρόεδρε, είναι διχασμένε. Εμεί είμαστε ενωμένοι στην θέση μα αυτή. Σα ευχαριστούμε πολύ. για την Ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Αριστερά και την Βόρεια Πράσινη Αριστερά. Ο κύριος Λότα Πίσκι παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπαρόζο, συνάδελφοι, και η δική μου ομάδα ενεργά συμμετείχε στις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων από κάποιους από αυτούς αποκομίσαμε μια οπωσδήποτε θετική εντύπωση. Λιγότερο ικανοποιημένοι είμαστε από κάποια χαρτοφυλάκια σε σχέση με την εκπροσώπησή τους. Αυτό αφορά και κάποιες ε, πιο ας το πω έτσι αδιαφανείς ε, ε, διεργασίες όσον αφορά την είπα το εκπρόσωπο των, για τα εξωτερικά όσον αφορά και το ταυτόχρονο αξίωμά της ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και αποδιαφήνιση αυτών των θεμάτων. Κάποιοι υποψήφοι μας απογοήτευσαν. Θα πρέπει να δούμε προς τα που θα, θα κινηθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια μέτρα είναι τα πιο σημαντικά για τους υποψήφιους ε, επιτρόπους. Σε αυτά τα ερωτήματα υπήρξαν γενικόλογες απαντήσεις και τέτοιες απαντήσεις που δεν μπορούν να υποστηριχθούν από εμάς. Παρόλη την αναφορά μιας κοινωνικής Ευρώπης με την απελευθέρωση και απορρίθμιση, με την ιδιωτικοποίηση ή με την έννοια flexicurity της ελαστικότητας και ασφάλειας συνεχίζουν κάποιοι να πορεύονται με αυτές τις έννοιες οι κοινωνικές ανάγκες των κοινωνικών συστημάτων βρίσκονται κάτω, άλλες προτεραιότητες ε, έχουν αντικαταστήσει αυτές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές, όμως δεν αλλάζει η πορεία από την εκμετάλλευση ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου. Και δεν βλέπουμε σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια και ε, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών τι πρέπει να γίνει. Ιδιαίτερα όσον αφορά και τα, τα, την πυρηνική ενέργεια και τα όπλα στην Ευρώπη. Κύριε Μπαρόζο, παρότι εκτιμούμε το ότι οι υποψήφοι από την ακρόαση αυτή παρουσιάστηκαν και έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Η δική μου ομάδα δεν μπορεί να εκφράσει θετική ψήφο στο Σώμα των Επιτρόπων. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματο της ομάδας Ευρώπη των Ελευθεριών και Δημοκρατιών, ο κύριος Νάτζελ Φάρατζ. Οι μελλοντικέ γενναίε, τα παιδιά, θα ακούνε μια ιστορία μια φορά και έναν καιρό η Ευρώπη ήταν διχασμένη, πόλεμος στα ανατολικά ήταν φτωχοί, είχαν τον κομμουνισμό που σκότωνε εκατομμύρια από τους πολί, των πολιτών του, αλλά ο τη της Εψίστης κατέρευσε το τείχος που τους χώρισε και 27 χώρες με 500 εκατομμύρια ανθρώπων μπόρεσαν να ζήσουν μαζί και εν ειρήνη. Όχι, όχι, συνεχίζεται η ιστορία. Ακούστε με, ακούστε με. Έχει κι άλλο. Ε, ας καθίσω τότε, μάλλον τέλειωσα. Πρώτη φορά είναι που με επικροτούν μέσα στο κοινοβούλιο τόσο πολύ και πραγματικά μπαίνω στον πειρασμό να καθίσω, να μην συνεχίσω την ομιλία μου. Αλλά πρέπει να συνεχίσω δυστυχώ, διότι συνεχίζεται το παραμύθι και ε, αυτοί που είχαν την εξουσία, οι πολιτικοί, ε, γίναν άπλιστοι, θέλανε τα λεφτά να τα κρατήσουν στην τσέπη του, θέλανε όλη την εξουσία, δεν θέλανε να παρετηθούν από τη δύναμη που είχαν και έτσι σκηνοθέτησαν το πιο θεαματικό γραφειοκρατικό πραξικόπημα οποιαδήποτε ιστορία και μάλιστα δεν χρειάστηκε καν το στρατό αυτό το πραξικόπημα, ήταν πολύ πιο ευφυή αυτή η πολιτική. Δημιούργησαν λοιπόν ένα σύστημα πολύ αποτελεσματικό που ονομαζόταν Συνθήκη της Λισαβόνα. και έτσι 27 άνθρωποι εξασφάλισαν απεριόριστη ανεφορίων εξουσία. Αυτοί εδώ, αυτοί εδώ ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να διατυπώσουν οποιοδήποτε νόμο θέλανε. Βεβαίω είχαν και τη σημαία του, βεβαίω είχαν και το εθνικό του το εθνικό τους ύμνο, αλλά προχωρήσαν ακόμα περισσότερο και θέλουν να φτιάξουν και κράτο, αγνώντα τη βούλη των λαών. Και έτσι ξαναδημιούργησαν, θέλοντα και εμεί, την, ε, τα δεινά του παρελθόντος, το σατανικό εκείνο σύστημα από το οποίο υπέφερε ο κόσμος στο παρελθόν. Και μάλιστα το αστείο σε όλα αυτά και το παράδοξο ήταν ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτή την ομάδα των 27 είχαν ήδη υπηρετήσει το σατανικό σύστημα του παρελθόντος. Και μάλιστα είχαν και ένα σύστημα νομισματικό το οποίο κατέρευσε, αλλά παρόλα αυτά δεν άκουγαν το λαό οι νέοι αυτοί οι αρχηγοί, οι νέοι αυτοί οι ηγέτες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά γίνανε και πιο σκληροί ακόμα και έτσι ρίξανε τόσα εκατομμύρια ανθρώπων στη φτώχεια, δεν τους άκουγαν καθόλου τους λαούς τους και έτσι χρειάστηκε οι λαοί τους να αντιδράσουν με τη βία για να ανακτήσουν τα, τα έθνη κράτη και τη δημοκρατία και το δίδαγμα από αυτό το παραμύθι είναι ότι δεν διδαχθήκανε τίποτε από την ιστορία. Και εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκεφτείτε πολύ καλά πριν τους δώσετε την εξουσία αυτή ότι υπάρχει το ιστορικό υπάρχει, έχει καταρρεύσει το σιδηρούν παραπέτασμα στην Ευρώπη, αλλά τώρα έχουμε μια νέα σιδηρά γροθιά, μια οικονομική σιδηρά γροθιά και δεν μπορούμε πάνω σε αυτήν. Ευχαριστώ πολύ, διακόπτει ο Πρόεδρος. σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Φάρατς, ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Głos zabierze pan Hans Peter Martin. Oh. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Χάνς Πέτερ Μάρτιν, παρακαλώ. Μετά από αυτό το παραμυθάκι που μόλις ακούσαμε, ας ξαναγυρίσουμε στην πραγματικότητα, θα έλεγα. Ο γιος μου είναι 17 ετών και μαθαίνει έντονα αγγλικά. Ε, Τα αγγλικά είναι γλώσσα εργασίας της Ευρώπης και ελπίζει ότι θα πάρει και μια καλή δουλειά. Ευρωπαίος, φιλοευρωπαίος, ε, πεπισμένα φιλοευρωπαίος. Έχει όμως ε, κορεστεί από τα όσα γίνονται στην ε, Ευρώπη και αναφέρονται και δημοσιεύματα τα οποία επιβαρύνουν την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, εκατομμύρια νέων Ευρωπαίων ελπίζουν ότι θα υπάρξει μια λειτουργούσα, τολμηρή δημοκρατία στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα. Τώρα, τι μα προσφέρεται από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Σώμα Επιτρόπων. Είναι οι ικανότεροι και οι καλύτεροι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται, αυτοί που χρειαζόμαστε. Είναι κάποιοι από κάποιου ε, υποψηφίου ε, που έχουν ε, ως αποτέλεσμα από πλευράς κάποιων ακροδεξιών όπως λένε να μην θεωρούμαστε εμείς ε, κομματική πολιτική κοινοβουλευτική ομάδα. Όμω είμαστε πεπισμένοι Ευρωπαίοι και θα θέλαμε να λειτουργήσουμε σωστά. Αν παίρναμε έναν βοηθό και θέλαμε να τον ε, ε, απασχολήσουμε θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να το κάνουμε. Πιθανότατα όχι. Για τι αρμοδιότητε από πλευρά Επιτρόπου τη Αυστρία σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο του από πλευρά ε, του Προέδρου υπάρχουν πραγματικά πολύ έμπειροι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι που θα μπορούσαν να να αναλάβουν έργο. Για παράδειγμα, γιατί δεν έχουμε τον Νότμα Κάρας ή κάποιον άλλον ανταυτών που προσφέρθηκαν. Γιατί δεν επιτρεπόταν. Διότι παρόλη τη συνθήκη τη Λισαβόνας είμαστε όμοιροι. Δεν είμαστε σε θέση αυτενεργά να λάβουμε αποφάσεις τελώς. Δυστυχώ, ε, και στο μέλλον δεν μπορούμε να επιλέξουμε έναν επίτροπο που θα τον καταψηφίσουμε ώστε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι του 19ου αιώνα, δεν είναι του 21ου και δεν είναι τολμηρό και δεν είναι αυτό το όραμά μα. Κρούω κινδύνου να μην συνεχίσουμε έτσι. Έτσι θα παίξετε το παιχνίδι των ε, ε, εθνικιστών. Ανταυτόν χρειαζόμαστε περισσότερη δημοκρατία όμω στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ για την δήλωσή σα, ε, λέει ο πρόεδρο. Ο Μπρούνο Γκόλνη τώρα που θα ήθελε να κάνει μια προσωπική δήλωση. 151. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακριβώς περί αυτού πρόκειται, θα είμαι πολύ σύντομος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Σούλτς, ε, οι υποψήφοι έχουν ε, ακριβώς προτείνει ανθρώπους, ε, έχουν προταθεί για... ωστόσο υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει αρνηθεί το αυτόμα. Αυτό έχει αναγνωριστεί και γι' αυτό και ήθελα να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η προφανής απόφαση της δικαιοδοσίας, της γαλλικής δικαιοδοσίας, δηλαδή το εφετείο, το κυρωτικό δικαστήριο, το οποίο έχει δώσει μια εξαιρετική απόφαση, ότι είχα διωχθεί με τη βάση τμήματων αποσπασμάτων φράσεων που είχαν ε, στοιχειοθετηθεί τεχνητά για να υπάρξει μια δήλωση και ακόμα και έτσι ε, ενώ διώχθηκα από τους πολιτικούς μου αντιπάλους αυτό δεν στάθηκε απέναντι στη δικαιοσύνη, απέναντι στον νόμο. Είναι μια πολύ σπάνια απόφαση διότι πρόκειται για μια ανακύρωση χωρίς ε, δικαίωμα παραπομπή σε μια άλλη δικαιοδοσία. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο από άποψη του Γαλλικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Αυτό έγινε για πρώτη φορά στην ε, ε, ε, ιστορία μας στην υπόθεση Dreyfus. Και κατά συνέπεια να προσθέσω ακόμα κάτι. Δεν είχα πει ότι η κυρία Άστον ήταν κομμουνίστρια, είχα πει ότι είχε αποτελέσει τμήμα αυτού του ειρηνισμού που ίσως ο Λένιν να είχε διακόπτει ο πρόεδρος, τον ομιλητή. Προσωπική δήλωση μόνο, κύριε γκόλνη, είπαμε. Σας ευχαριστώ. Πάνιε Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκόλνης. Προσωπική δήλωση αποκλειστικά είχαμε αναφέρει. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία έχουμε όλη συνείδηση της σημασίας της ψηφοφορίας αυτής. Έχουμε λοιπόν στην ημέρηση διάταξη την ψηφοφορία για τρεις προτάσεις ψηφισμάτων ως προς την έγκριση της Επιτροπής Συλλογικού Οργάνου. Προχωρούμε στην ψηφοφορία της προτάσεως ψηφίσματος των πρασίνων, χωρίς τροπολογίες. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνούμε τώρα στην ψηφοφορία της προτάσεως ψηφίσματος της Νομοσπονδιακής Ομάδας Αριστεράς ε, Πράσινων Σκανδιναβών υπέρ, χωρίς ψηφοπολογίες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνούμε στην ψηφοφορία του προτάσματος ψηφίσματος της ομάδας των Ευρωπαίων Ταριθμιστών και Δημοκρατών χωρίς τροπολογίες με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία.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 Στην ημερήσια διάταξη προβλέπεται τώρα η ψηφοφορία για μια πρόταση ε, αποφάσεως για τη νέα σύνθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ψηφίζουμε το σύνολο της αποφάσεως, προτάσεως αποφάσεως με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εψήφισαν υπέρ 488, 137 κατά, 72 αποχές. Σας ευχαριστώ. I would like... Και τώρα θα ήθελα να εκφράσω θερμά συγχαρητήρια στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Συλλογικό Σώμα και τον Πρόεδρο Μπαρόσο. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Πολλή δουλειά σας περιμένει, μας περιμένει. Πολλές είναι οι προσδοκίες των πολιτών μας, υψηλέ οι προσδοκίες των πολιτών μας. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε τη δουλειά και να φέρουμε τα αποτελέσματα. Και καλό αμέσως τον πρόεδρο της εναλλασσομένης προεδρίας και τον, τον κύριο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ενημερωθούν, θα τους ενημερώσω μάλλον αμέσως για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για να αναλάβει τα καθήκοντά της Νέα Επιτροπή μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2014. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Uh, yes, colleagues. Uh, I didn't know about that. Well, you, you take the floor, yeah? Okay. Uh, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ να καθίσετε, διότι ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου θα ήθελε να μας πει δύο λόγια. Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Why I didn't know about that. Uh, Statement by the Council. Δήλωση του Συμβουλίου, παρακαλώ. Secretary of Chair. Well. Uh, ε, Mr. President Barroso. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, Δύο λεπτά παρακαλώ. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ σύντομα να εκφράσω την ικανοποίησή μας από πλευράς του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συγχαρώ τον κύριο Μπαρόζο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της για την ψήφο εμπιστοσύνη τη οποία έτυχε και την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τη οποία απέλαβαν από το σώμα την Ευρωβουλή τους επόμενου μήνε και χρόνια στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτά τα δύο θεσμικά όργανα θα διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκλήσεις της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, πρόκληση της ασφάλειας, της παγκοσμιοποίησης, οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Το να αποφύγουμε μια κρίση σαν αυτήν την οποία, στην οποία βρισκόμαστε ακόμα, την εκκίνηση των νέων πρωτοβουλειών από πλευρά των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την συνθήκη τη Λισαβόνα, την πρωτοβουλία, ανάληψη πρωτοβουλία των πολιτών, την ρήτρα αλληλεγγύη και φυσικά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων, διπλωματική υπηρεσία και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και εμεί ω Συμβούλιο ευχόμαστε και επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση αυτή τη δύναμη να εργαστεί. Σίγουρα έχει πολλέ εξουσίες, όχι απεριόριστες όπως προαναφέρθηκε, αλλά έχει εξουσίες για να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστεί γοργά και αποτελεσματικά, διότι οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν και εύχονται να εργαστεί έτσι αποτελεσματικά και, και γοργά. Και άμεσα μετά από αυτή την περίοδο αβεβαιότητας, θεσμικής αβεβαιότητας που πέρασε η Ευρώπη, να μπορέσουμε όλοι μας να εργαστούμε, να ξανακερδίσουμε το χαμένο χρόνο και να δρομολογήσουμε αμέσως αυτή την πολιτική, νέα πολιτική φάση, αυτή τη νέα κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, δηλαδή να περάσουμε τελεσίδικα και καθοριστικά στον 21ο αιώνα Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω κύριε Μπαρόζο για τον ευρωπαϊκό λόγο που έχετε διατυπώσει ότι θα έχετε κάθε συνεργασία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα έχετε τη συνεργασία του Συμβουλίου όπως απαιτείται για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη και να προσεγγίσουν περισσότερο οι ε, πολίτες που εκπροσωπούνται από αυτή την Ευρωβουλή να μπορέσουν οι πολίτες αυτοί να βρεθούν στον πυρήνα, στην καρδιά της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Υφυπουργό για τα Ευρωπαϊκά Θέματα της Ισπανίας, εκ μέρους του Συμβουλίου, κύριο Καρίγιο. Κύριε Μπαρόσο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σύντομα θέλω να εκφράσω εξ ονόματός μου αλλά και εξ ονόματος όλων των ε, επιτρόπων την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μόλις ε, μας ε, δείξατε και είμαι περήφανος για την, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας γιατί βλέπω πως υπάρχει ισχυρή στήριξη από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρώπη ε, να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για τα θερμά του λόγια. Πιστεύω πως είμαστε τώρα σε θέση να στρωθούμε στη δουλειά. Αλλά θα ήθελα να σχολιάσω μόνο το εξή. Κατά τη διάρκεια αυτής της ψηφοφορίας άκουσα εδώ κάποιες παρατηρήσεις και θέλω σαφώς και ξεκάθαρα να πω πως ε, όσοι συγκρίνουν ε, την απολυταρχική Σοβιετική Ένωση με την Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρουν καν τι θα πει να ζήσει κανείς σε δεκτατορικό καθεστώς και δεν ξέρουν τι θα πει δημοκρατία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι δημοκρατία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εκλεγμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από εσά που είστε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών τη Ευρώπη. Αυτό είναι δημοκρατία. Και πιστεύουμε πω τώρα με τη δημοκρατική αυτή νομιμότητα που μα δώσατε, που μα δώσατε εσείς ορίζοντας ε, υπερψηφίζοντας τους υποψήφιους των 27 δημοκρατικό εκλεγμένων κυβερνήσεων είμαστε σε θέση να δουλέψουμε για τη δημοκρατία και για την Ευρώπη, την Ευρώπη που είναι ένας φάρος ελευθερίας για ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε έτσι αυτό το σημείο τη ημερήσια συνέντευξη και είναι και η κατάλληλη στιγμή για να δώσουμε συγχαρητήρια.